ισχύουν εξίσου για το 2012 και το 2013. Είναι η ίδια διαδικασία. Τώρα έχω την επόμενη ανακοίνωση. Ο κ. Τζο Higgins και ο κ. Άλαν Κέβιν με ενημέρωσαν ε, γραπτός για την εκπνοή της ε, θητείας τους ως ευρωβουλευτές λόγω του ότι εξελέγησαν στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται αυτές τις πληροφορίες και σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του εσωτερικού κανονισμού που αφορά την εκλογή Ευρωβουλευτού ε, σε Εθνικό Κοινοβούλιο στις εκλογές δηλώνει ότι αυτές οι δύο έδρες είναι κενές από τις 25 Φεβρουαρίου ε, ενεστώτος έτους. Και τελευταία ανακοίνωση, η υπογραφή των νομικών πράξεων γίνεται, λαμβάνει η χώρα μέσα της κανονικής, της συνηθισμένης διαδικασίας. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου και τη Δευτέρα θα